Τη ουσία. Άλλη ανακοίνωση, όπω θα θυμάστε, στις 13 Δεκεμβρίου 2016, ο πρόεδρος επέβαλε μια ακύρωση στον κύριο Βόιτ, που είχε παραβιάσει την υποχρέωση κοινοποίηση ε, σύμφωνα με τον κώδικα διοντολογία και τα μέτρα εφαρμογή του. Στι 27 Δεκεμβρίου, ο κύριο Βόιτ υπέβαλε ε, προσφυγή προς την, ε, εναντίον αυτή τη απόφαση. Τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου, το Προεδρείο εξέτασε την προσφυγή και επιβεβαίωσε ομόφωνα την απόφαση του Προέδρου να επιβάλλει μια προειδοποίηση προς τον κύριο Βόιτ.